arrêtavano. Questo. May I um, try to give you some practical advice, uh, please? Λοιπόν, να δούμε κάποια πρακτικά θέματα. Με ακούτε, ακούμε ελληνικά. Στο 7 ακούμε. Ωραία, ακούμε έτσι. Μπράβο, τέλεια. Λοιπόν, μισό λεπτό σταματάω, σταματάω να μιλάω εξηγεί εξηγή, για τα κανάλια για να αλλάξω ακουστικά γιατί δεν έχω καλά ακουστικά και το ξανανοίγω, μην τρομοκρατηθείτε. So, until the discussion we have with all of us, please don't press the button to speak. And uh, we will see later on Uh, how to do it. I hope that... Ωραία. Εντάξει, έτσι. Λοιπόν, λέει ο κύριος ότι έχουμε διερμηνία όλοι στη γλώσσα μας και βέβαια ε, τα κανάλια σας ε, τα έχετε βρει. Όσοι λοιπόν χρειάζεστε διερμηνία, Μπορείτε να σηκώσετε τα χέρια σας, λέει, αν με ακούτε μέσω της διερμηνίας. Ναι, αν ακούτε, δηλαδή αν δεν έχετε πρόβλημα με τα κανάλια, σηκώστε το χέρι σας. Οι, οι, κυρίες οι υπόλοιπες έχουν, με ακούνε. Ναι. Με ακούτε έτσι όλες, ωραία, εντάξει. Ωραία. Αν κάποιος έχει πρόβλημα και δεν ακούει, αν και δεν βλέπω κανένα να παραπονιέται, ωραία, μάλλον όλοι είμαστε εντάξει, λοιπόν, λέει ο συντονιστής. Καταρχάς, πριν ξεκινήσουμε, ο πρόεδρος της ημέρας, ο Χωσέ Μανουέλ Φρέσνο, δυστυχώς δεν θα μπορέσει να έρθει ανάμεσά μας για την ώρα, διότι έρχεται από την Ισπανία και είχε καθυστέρηση. Έρχεται μέσω Παρισιού και τον αναμένουμε γύρω στις 11 λόγω της καθυστέρησης. Ωστόσο, εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε και βεβαίως ε, θα τον αντικαταστήσω εγώ. Εγώ είμαι ο Λούντο Χόρεμανς, είμαι ο πρόεδρος ε, του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Φτώχειας. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ προκειμένου να αντικαταστήσω τον Χωσέ Μανουέλ Φρέσνου, πράγμα το οποίο είναι κάτι πολύ δύσκολο. Ε, πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη και από τον κύριο, να ζητήσουμε συγγνώμη, μάλλον μας ζητάει συγγνώμη και ο κύριος Άντορ, ο Επίτροπος, γιατί δεν μπόρεσε να είναι ανάμεσά μας και θα αντικατασταθεί. Τώρα θέλω να καλωσορίσω και την κυρία Πέρεθ, η οποία είναι η πρόεδρος της ε, Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και ένα ιδιαίτερο καλωσόρισμα στην κυρία Μαρτίνεθ, η οποία εκπροσωπεί την Ισπανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία διοργανώνει την ευρωπαϊκή μας συνάντηση και είμαστε ευγνώμονες βεβαίως γι' αυτό, επειδή η κυβέρνησή σας ως προ... πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εξάμεινο μέχρι το Δεκέμβριο αποφάσισε να διοργανώσει την Ευρωπαϊκή Συνάντηση όπως κάνουν και όλες οι προεδρίες κάθε χρόνο. Θέλω να καλωσορίσω επίσης ε, και τον... την πρόεδρο της Κοινωνικής Επιτροπής που είναι μαζί μας και ένα καλωσόρισμα στην κυρία Αδέλια Φερνάντεθ, η οποία εκπροσωπεί την προηγούμενη Ευρωπαϊκή Συνάντηση, την 8η δηλαδή, και η οποία βεβαίως θα μας καταθέσει τη μαρτυρία της. Λοιπόν, τούτου λεχθέντος και αφού έχω παρουσιάσει όλους τους εξέχοντες καλεσμένους, θα γίνει και μια σύντομη εισαγωγή από όλους τους ε, προσκεκλημένους και γι' αυτό θέλω να ε, πρώτα να καλωσορίσω όλες τις αντιπροσωπίες από την κάθε χώρα και θα περάσω γρήγορα τη λίστα των αντιπροσωπιών και όταν θα μιλάω για την κάθε χώρα αν θέλετε σηκωθείτε η κάθε αντιπροσωπεία όταν θα φτάνω στη σειρά τη, έτσι ώστε να δούμε ότι είστε παρόντες εδώ στην ένατη Ευρωπαϊκή ε, Συνεδρίαση για τους ανθρώπους που βιώνουν τη φτώχεια. Ξεκινάω λοιπόν με την Αυστρία. Αυστριακή αντιπροσωπεία, σηκωθείτε. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε. Βέλγιο, βελγική αντιπροσωπεία παρακαλώ. Καλώς ήρθατε. Βουλγαρία παρακαλώ. Καλώς ήρθατε Βουλγαρία. Η Τσεχία. Καλώς ορίσατε. Η Κύπρος παρακαλώ. Καλώς ήρθατε Κύπρο. Η Δανία. Καλώς ήρθατε Δανία. Η Εστονία παρακαλώ. Καλώς ορίσατε. Η Φινλανδία. Η Γαλλία. Καλώς ήρθατε Γαλλία. Η Γερμανία. Η Ελλάδα παρακαλώ. Καλώς ήρθε η Ελλάδα. Η Ουγγαρία. Η Ιρλανδία. Η Ιταλία. Η Λετωνία. Η Λιθουανία. Καλωσορίσατε. Το Λουξεμβούργο. Η Μάλτα. Οι κάτω χώρες. Νορβηγία. Η Πολωνία. Πορτογαλία. η Ρουμανία η Σλοβακία η Σλοβενία η Ισπανία Καλώς ήρθατε. Η Σουηδία. Το Ενωμένο Βασίλειο. Και νομίζω ότι κάναμε το γύρο όλων των αντιπροσωπιών. Καλωσορίσατε λοιπόν κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη συνεδρίαση διοργανώνεται από την Ισπανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αντιπροσωπείες όμως είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που είναι το επίκεντρο της συνεδρίασης. Προσκαλούμε εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων, των Εθνικών Κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χαιρόμαστε πάρα πολύ που κάθε φορά η εκάστοτε Προεδρία θέλει να διοργανώνει την Ευρωπαϊκή μας συνεδρίαση. Θα προσπαθήσω να δώσω, αν θέλετε, κάποια μεγαλύτερη ορατότητα στις ομάδες των προσκεκλημένων μας να φανούν λίγο περισσότερο και επειδή βρισκόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλω να ζητήσω από τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου παρόντα εδώ να σηκωθούν παρακαλώ. Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρακαλώ σηκωθείτε. Καλωσορίσατε. Και η βοηθή των μελών, παρακαλώ. Η βοηθή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Ευρωβουλευτών. Όσοι έχετε έρθει, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και εσάς. Καλώς Θα θέλαμε τώρα να ζητήσουμε από τους ανθρώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σηκωθούν για να τους καλωσορίσουμε και αυτούς. Όσοι είστε εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Διοίκησης, παρακαλώ σηκωθείτε. Θέλουμε να σας καλωσορίσουμε και εσάς. Και θέλω να ζητήσω και από τους υπόλοιπους εκπροσώπους των εθνικών κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σηκωθούν, έτσι ώστε να σας καλωσορίσουμε. Όλοι οι εκπρόσωποι των ε, κυβερνήσεων, των διοικήσεων, σηκωθείτε παρακαλώ. Καλωσορίσατε και ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Και υπάρχουν και άλλοι προσκεκλημένοι, ίσως που δεν ανήκουν σε καμία από αυτές τις κατηγορίες. Άνθρωποι από μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ας πούμε, και από άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Μπορείτε παρακαλώ να σηκωθείτε. Μη κυβερνητικέ οργανώσεις, Οργανώσεις κοινωνία των πολιτών, παρακαλώ. Ωραία. Έρχονται, έρχονται, έρχονται. Να τι σηκώνονται, αυξάνονται και πληθύνονται. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Τώρα, αν έχω παραλείψει κάποιον, από οποιαδήποτε κατηγορία, παρακαλώ να σηκωθείτε. Ή είμαστε όλοι εντάξει. Α, ο κύριος. Καλώς ορίσατε. Ωραία. Λοιπόν, κατόπιν των ε, συστάσεων, νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι βρισκόμαστε ήδη στην ένατη Ευρωπαϊκή Συνεδρίαση και στον, στην ένατη χρονιά καταπολέμησης της φτώχειας. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ευκαιρία που έχουμε να συναντηθούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το όργανο το οποίο εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαιρόμαστε ιδιαίτερα και είμαστε ευγνώμονες διότι και Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ισπανική Προεδρία μας διοργάνωσαν αυτή μας την Ευρωπαϊκή Συνεδρίαση. Ε, το γνωρίζουμε ήδη, αλλά θα σας το ξαναπώ. Είναι μια πολύ σημαντική συνεδρίαση συγκεκριμένη. Όχι μόνο επειδή βρισκόμαστε στο Ευρωπαϊκό Έτος πολέμηση της Στόχιας, αλλά επειδή ταυτόχρονα θέλουμε να δώσουμε περισσότερες απαντήσεις σε όλες τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει σε προηγούμενες ευρωπαϊκές συνεδριάσεις. Και έχουμε έναν μακρύ κατάλογο προτάσεων. Και τον έχουμε παρουσιάσει και στις κυβερνήσεις και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα λάβουμε κάποιες απαντήσεις. Ακόμη και όταν η απάντηση δεν είναι ακριβής και λέει ότι δεν ξέρουμε πώς να εφαρμόσουμε το τάδε ή το δίνα. Παρ' όλα αυτά δίνει βάση για συζήτηση και τα εργαστήρια που, στα οποία θα χωριστούμε μετά την Ολομέλεια ακριβώς θα επεξεργαστούν αυτά τα θέματα. Αφού θα ακούσουμε λοιπόν τους ομιλητές μας, μετά θα χωριστούμε στα, α, στις ομάδες. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική συνεδρίαση. Η φωνή και οι προτάσεις των ανθρώπων που ήδη βιώνουν προβλήματα είναι πολύ σημαντικά πράγματα να ακούγονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο όπως και στο εθνικό. Όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι σε εθνικό επίπεδο έχουν και πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Συμβούλιο των Υπουργών λαμβάνει πολύ συχνά αποφάσεις. Είναι οι εκπρόσωποι των εκάστοτε κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί αποφασίζουν ε, για τις προτάσεις. Προσμονούμε λοιπόν να ακούσουμε προτάσεις και να συζητήσουμε το πώς μπορούν να υλοποιηθούν οι συγκεκριμένες προτάσεις ή να συζητήσουμε τα προβλήματα. Γι' αυτό πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό στόχο που έχει θέσει η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Να καταφέρουμε να συνεχίσουμε και στο μέλλον τη δουλειά μας. Ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντική στιγμή η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική, η Ευρώπη 2020, όπως τη λέμε, Europe 2020, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, οι υπεύθυνοι των ευρωπαϊκών θεσμών, την περασμένη εβδομάδα έλαβαν απόφαση σχετικά με τους μεγαλεπίβολους στόχους που αφορούν ε, τη στρατηγική και την ένταξη προκειμένου να γίνει ένα πρώτο βήμα για την εξάλληψη της φτώχειας. Διότι αυτό θα πρέπει να αποτελεί τον απότερο σκοπό για όλους μας. Η απόλυτη εξολόθρευση της φτώχειας που αποτελεί ντροπή για μια τόσο ευήμερη περιφέρεια όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε λοιπόν μετά την απόφαση που ελήφθη την περασμένη εβδομάδα να συνεχίσουμε περαιτέρω και να υλοποιήσουμε αυτά που ανακοινώθηκαν. Τώρα θα δώσω το λόγο στους ε, εισηγητέ μας και καταρχάς, ε, επειδή βρισκόμαστε τόσοι άλλους εδώ, καλεσμένοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα δώσω το λόγο στην κυρία, στην κυρία Περέσα, η οποία είναι η πρόεδρος της Επιτροπής για την Απασχόληση και των Κοινωνικών Υποθέσεων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή που κάνατε και για την παρουσίαση που κάνατε για όλους εμάς. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μάλλον είναι ασυνήθιστη μια τέτοια πρακτική και πραγματικά χαιρετίζω αυτή την πρωτοτυπία που μας δίνει την δυνατότητα να συνεργαστούμε επικοδομητικά αυτές τις μέρες. Καλωσορίσατε λοιπόν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι είναι η πρώτη φορά που λαμβάνει η χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά εδώ πρόκειται για τον οίκο όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Συνεπώς η δουλειά που κάνετε όλοι μαζί, το έργο που παράγετε, προκειμένου να ακουστεί η φωνή αυτών που δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα, αυτών που δεν ακούγεται ακριβά, ακριβώς η φωνή τους και όπως πρέπει, Χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχουν τόσοι πολλοί συνάδελφοι εδώ, οι οποίοι εκπροσωπούν διαφορετικά όργανα και θεσμούς και που είναι παρόντες εδώ για να σας ακούσουν, να μάθουν από σας και να μάθουν να δουλεύουν καλύτερα λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες και προβληματισμούς σας. Το είπατε κι εσείς. Η διάσκεψη λαμβάνει χώρα σε μια στιγμή αγώνα. Διότι γνωρίζετε, αυτή η στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2020, δηλαδή η στρατηγική για την καταπολέμηση, την εξάλληψη της στόχης και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, δεν ήταν κάτι κεκτημένο. Ακόμη και αυτή τη χρονιά που διανύουμε, που είναι η χρονιά καταπολέμησης στόχης και κοινωνικού αποκλεισμού. Γι' αυτό και χαιρετίζω την κινητοποίησή σας και την αποφασιστικότητά σας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ισπανικής Προεδρίας και όλων των συναδέλφων που βοήθησαν να κερδίσουμε αυτή τη μάχη, διότι από τούτο και στο εξής ο στόχος της εξάλληψης της στόχιας εγγράφεται στην ατζέντα των, ε, των αρχικών κρατών και κυβερνήσεων. Είναι λοιπόν μια πρώτη μάχη που κερδίσαμε όλοι μαζί και θεωρώ ότι τώρα πρέπει να προχωρήσουμε βάσει αυτής της απόφασης. Ξέρετε, ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι καμιά φορά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Τι είναι η φτώχεια, πώς τη μετράμε, πώς την καταπολεμούμε. Έχουμε την αίσθηση ότι είναι μια παλιά ιστορία. Ωστόσο, είναι πάντα πάνω στο τραπέζι. Γι' αυτό Πρέπει διαρκώς να βρίσκουμε νέα μέτρα, νέα εργαλεία καταπολέμησής της. Και ε, επ' αυτού θα εκφραστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όμως υπολογίζω ότι σε αυτή την περίοδο κρίσης που διανύουμε, η κρίση επηρεάζει αυτούς που έχουν μετοχές, έτσι, γιατί από εκεί γεννιέται. Αλλά δεν επηρεάζει μόνο αυτού, επηρεάζει και τους στοχότερους και οι συνέπειε μια τέτοια ε, κρίση, την οποία βιώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει συνέπειε στην ανακατανομή. Όχι ανακατανομή όπως αυτή που επιθυμούμε συχνά, αλλά έχει ανακατανομή αρνητικών συνεπειών. Και βρισκόμαστε σε μια στιγμή όπου βλέπουμε πολύ καλά. Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται βάσει των υποχρεώσεων που έθεσαν οι αγορές προκειμένου να μειώσουν τον προϋπολογισμό τους. Και πολύ φοβούμε και όλοι θα πρέπει να φοβόμαστε ότι αυτή η μείωση του προϋπολογισμού βασικά καταρχάς θα μειώσει τον προπολογισμό τον οποίο εμείς χρειαζόμαστε προκειμένου να κερδίσουμε τη μάχη της καταπολέμησης της στόχιας. Το πρώτο παράδειγμα προφανώς, και το έχω σημειώσει ότι αποτελεί και πρότασή σας, έτσι, η περσινή σας πρόταση. Λοιπόν, πρόκειται για το θέμα της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες. Φυσικά, υπάρχει ο τρόπος με τους οποίους οι πιο φτωχοί ε, έχουν πρόσβαση. Δηλαδή, πώς ασκούν αυτό τους το δικαίωμα. Πώς ένα ε, φτωχό παιδάκι θα πάει στο σχολείο πώς ένα ε, φτωχό παιδάκι δεν θα εγκαταλειφθεί από το σχολικό σύστημα. Υπάρχει όμως και το θέμα του πώς η εκπαίδευση, η παιδεία χρηματοδοτείται. Πώς το σύστημα υγείας χρηματοδοτείται και σε αυτή την ε, περίοδο εδραίωσης των προπολογισμών από τα κράτη-μέλη πρέπει να διαβάσουμε ένα πολύ δυνατό μήνυμα για να πούμε ότι ο βασικός μας πλούτος προκειμένου να εξέλθουμε από την κρίση είναι ακριβώς να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, να φροντίσουμε έτσι ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση στις πλούσιες κοινωνίες που γνωρίζουμε στην Ευρώπη. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, θέλω απλώς ε, να σας πω εξ ονόματος όλων των συναδέλφων μου της Επιτροπής ε, Κοινωνικών Υποθέσεων ότι δεσμευόμαστε να αγωνιστούμε και θέλω επίσης να αντιδράσω πάνω σε δύο-τρία σημεία των συμπερασμάτων σας της ε, περσινής συνεδρίασης. Θέτησε χθε την έκθεση της συναδέλφου που θα παρέμβει κάποια στιγμή, η οποία κάνει μια εξαιρετική δουλειά, προκειμένου να εντοπίσει πως το θέμα του ελάχιστου εισοδήματο είναι στοιχείο κλειδί στη στρατηγική καταπολέμηση της φτώχειας. Είναι πολύ δύσκολος ο αγώνας αυτός, χρειαζόμαστε την υποστήριξη της Προεδρίας προκειμένου να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Νομίζω όμως ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε αυτή την έκθεση που είναι κάτι πολύ σημαντικό τώρα πια. Κατόπιν, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους θα πραγματοποιήσουμε διάφορες εκδηλώσεις βάσει αυτής της ε, δέσμευσης. Έχουμε, ξέρετε και στις 19 Οκτωβρίου, μια συνεδρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επίσημη συνεδρίαση, όπου διάφοροι θύνοντες θα έρθουν να μιλήσουν. Και τώρα δύο-τρία λόγια όσον αφορά τα συμπεράσματά σας της περσινής χρονιάς. Το είχατε πει και πέρσι. Οι κίνδυνοι πολλών ε, ζημιών από είναι εξαιτία της κρίση, είναι ένα θέμα επίκαιρο. Είναι κάτι που στο Ευρωκοινοβούλιο το υπολογίζουμε, το μετράμε. Μεταξύ των Υπουργών μερικές φορές υπάρχουν κάποιες ανισορροπίες όσον αφορά αυτά που λέγονται μεταξύ ας πούμε των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και των Υπουργών Κοινωνικών Υποθέσεων. Μερικές φορές η ζυγαριά γέρνει κάπως δυσανάλογα. Άρα πρέπει να αγωνιστούμε προκειμένου οι Υπουργοί Κοινωνικών Υποθέσεων όταν μεταφέρουν χρήσιμα μηνύματα, συνήθως έτσι γίνεται, να εισακούγονται από τους υπουργού Οικονομικών. Και η διάφορη ανα, αναθεώρηση των λογαριασμών, η αναθεώρηση των χρεών, των κρατών, να μην ε, μεταφράζεται μέσα από την κατάρριξη και την καταστροφή των κοινωνικών μας μοντέλων. Όσον αφορά το θέμα δικαιώματος στη στέγαση, θεωρώ ότι ε, εμείς την καταπολέμηση της στόχης το γνωρίζουμε πολύ καλά. Είναι δύσκολη άσκηση αυτού του δικαιώματος. Η στέγη, η υγεία, η παιδεία. Τα γνωρίζουμε καλά, γι' αυτό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν θα δούμε ποιοι είναι οι διάφοροι δείκτες, πώς δηλαδή, εντάξει, είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα μειώσουμε τη φτώχεια. Ωραία. Πρέπει να το επιβλέψουμε. Πώς τη μειώνουμε δηλαδή τη φτώχεια. Στα πλαίσια αυτής της ε, επιτήρησης, αν πράγματι υπάρχει καταπολέμηση, για μας ε, το να ασχοληθούμε με το πώς λύνουμε τα προβλήματα των αστέγων είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Είναι ένα θέμα που αναδύεται συχνά και που πρέπει να μας απασχολεί. Σας είπα, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Μίλησα ήδη για την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. Απλώς θέλω να σας πω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ έχω την ευθύνη μιας έκθεσης της αξιολόγησης της κρίσης και στην έκθεση αυτή ζητώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε έναν απολογισμό των συνεπειών της κρίσης στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, διότι έτσι θα μπορέσουμε να επανακινητοποιήσουμε ε, το σύστημα για να ε, βελτιώσουμε πάλι τις κοινωνικές υπηρεσίες και να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις βεβαίως. Ε, πέρσι μιλήσατε επίσης και τονίσατε το θέμα της πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Μια έτσι παγκόσμια πρόσβαση και πρέπει να σας πω ότι είναι ένα από τα σημεία των συμπερασμάτων μιας πρότασης που έγινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον κύριο Μάριο Μόντι, τον οποίο είχαμε ανάμεσά μας στην Γενική Διεύθυνση πριν από δύο μέρες. Εμείς είναι κάτι το οποίο το υποστηρίζουμε, έτσι, την πρόσβαση στο τραπεζικό λογαριασμό. Τελευταίο σημείο, το ανέφερα ήδη, είναι το ελάχιστο εισόδημα με βάση πάντα την ε, εισήγησε τη συναδέλφου είναι ένα σημείο το, στο οποίο θα μας βρείτε δίπλα σας. Αυτές οι διεκδικήσεις τις δικές σας θα τις μεταφέρουμε και εμείς παραπέρα. Δεν ήθελα να μακρηγορήσω άλλο, θέλω να σας ευχηθώ επιτυχία στις εργασίες σας και καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και να σας πω ότι για μας, τους Ευρωπαίους νομοθέτες, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε επαφή μαζί σας και εσείς να μας βοηθάτε να γινόμαστε καλύτεροι νομοθέτες στην υπηρεσία όλων όσων μοιραζόμαστε, όπως είναι η καταπολέμηση της φτώχειας. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστούμε την κυρία Έρες για τις πρώτες απαντήσεις που δώσατε σχετικά με αυτά τα πάρα πολλά σημαντικά ζητήματα για τους ανθρώπους που βιώνουν τη φτώχεια και πράγματι αυτή η προσπάθεια, αυτός ο αγώνας σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει Πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά για να επηρεάσουμε την πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πολιτική που σχετίζεται στην αντιμετώπιση της φτώχειας, της εξάπλωσης της φτώχειας, γιατί ξέρετε, παντού ακούμε για μέτρα λιτότητας, αλλά αυτά τα μέτρα λιτότητας δυστυχώς πλήττουν περισσότερο τους ευάλωτους και κυρίως αγγίζουν τις λεγόμενες κοινωνικές δαπάνες. Και οι κοινωνικές δαπάνες, όπως πολύ σωστά το είπατε, επί της είναι επενδύσεις και δεν πρέπει αυτές τις δαπάνες, κοινωνικές δαπάνες να τις βλέπουμε σαν κόστη. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία η ε, Μαρτίν, Μαρτίνες, Ιζαμπέλα Μαρτίνες, εκπροσωπεί την Ισπανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. πολύ. Ε...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 Καλώς ήρθατε λοιπόν όλοι σε αυτό το χώρο της συμμετοχής που έχει βεβαίως ε, και περιφερειακή και εθνική εμβέλεια. Η δική σας γνώμη είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να ε, κρίνουμε την πραγματική εμβέλεια των πρωτοβολιών που υποτίθεται ότι βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσής μας. Αυτή η συμβολή με τις μαρτυρίες προσωπικών εμπειριών Πραγματικά εμφανίστηκε πάρα πολύ και στη διάσκεψη και στην εναρκτήρια διάσκεψη που έγινε τον Ιανουάριο που μας πέρασε στην Ισπανία, στη Μαδρίτη. Σήμερα είμαστε πεπισμένοι ότι μόνο μέσω αυτής της μεθόδου ε, ε, μπορούμε πραγματικά να αξιολογήσουμε με βεβαιότητα εάν οι πολιτικές καταπολέμησης της ε, φτώχειας είναι χρήσιμες και κατευθύνονται στη σωστή κατεύθυνση. Για το λόγο αυτό, σε αυτή τη νέα συνάντηση θέλουμε να πάμε ακόμη πιο πέρα από τις άλλες περιπτώσεις και θέλουμε να το κάνουμε βάσει τριών γραμμών ε, κεντρικών. Σε πρώτη φάση θέλουμε να συζητήσουμε πραγματικά πού έχουν οδηγήσει οι προηγούμενες οκτώ συνεδριάσεις. Να, να δούμε τον αντίκτυπο που είχαν αυτές οι συνεδριάσεις στα άτομα που βιώνουν τη φτώχεια, καθώς και τι πολιτικές ε, αποφάσεις έχουν ληφθεί. Σε δεύτερη φάση θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων των οργανώσεων και των ευρωπαϊκών θεσμών και τέλος, μέσα από την ανάλυση και τη συζήτηση, θα... Οι αντιπροσωπείες των ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια θα παρουσιάσουν ένα σχέδιο δράσης προς ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των επόμενων δέκα ετών. Αυτό πραγματικά είναι το σημαντικό. Να δημιουργηθεί ένα σχέδιο το οποίο θα μας οδηγήσει, το οποίο θα μας ε, τοποθετήσει εκ νέου στις κοινωνικές οργανώσεις και στα κράτη-μέλη ε, μπροστά από μια ευθύνη να λειτουργήσουμε συγκεκριμένα με συγκεκριμένους στόχου που θα φτάσουν στην καρδιά των ανθρώπων που πιο πολύ χρειάζονται. Υπ' αυτή την έννοια η, η Ισπανία θέλει να δεσμευτεί και να προωθήσει την ένταξη αυτού του κοινωνικού σχεδίου δράσης στην τελική διακήρυξη που θα γίνει στο, Ευρω... στο τέλος του Ευρωπαϊκού Έτου Καταπολέμησης της Στόχης και Κοινωνικού Αποκλεισμού το 2010. Αυτό το έγγραφο θα το εκπονήσουμε από κοινού με το Βέλγιο μέσα στα επόμενα εξάμηνα. Θέλουμε η καταπολέμηση της στόχιας να αποτελέσει έναν ε, σημαντικό στόχο έτσι ώστε όλοι να ε, συμμετέχουμε. Είναι μία από τις προτεραιότητες που έθεσε η Ισπανία κατά τη διάρκεια της ε, προεδρίας της. Και τα αποτελέσματα βεβαίω θα συνεχιστούν και μετά την Προεδρία. Η Ισπανία προσπάθησε να ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα έτσι, πολύ μεγάλο επίβολο. Μας ενδιαφέρει να το θέσουμε το θέμα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ατζέντας αυτούς τους μήνες. Έχουμε εργαστεί προκειμένου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές να μην χάσουμε την προοπτική ε, του τι σημαίνει κοινωνικό ευρωπαϊκό μοντέλο. Πράγμα που μας ε, επέτρεψε να δείξουμε ένα καλύτερο πρόσωπο στον κόσμο. Μας ενδιαφέρει η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού για να μοιραστούμε καλές πρακτικές και να διευρύνουμε τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες όσον αφορά τα μέτρα προστασίας. Υπό τις παρούσες συνθήκες που βεβαίως ε, τονίζονται από την οικονομική κρίση, η Ισπανία μίλησε για μια εδραίωση και μια προσπάθεια των κοινωνικών πολιτικών στην ευρωπαϊκή ε, ε, σκηνή προκειμένου να βοηθήσει τους πιο ευαίσθητους και να εγγυηθεί κάποια ελάχιστα μέτρα για την καλή τους διαβίωση. Οι πρώτες μας προτάσεις έγιναν ήδη τον Ιανουάριο κατά τη διεθνή, την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη και μας ενδιαφέρει να κάνουμε πιο εύκολη τη λήψη αποφάσεων. Με τον ίδιο σκοπό τον ε, Απρίλιο είχαμε μια Ευρωπαϊκή Σύνοδο στην Κόρδοβα που αφορούσε ακριβώ του πιο εύθραυστου ε, και κοινωνικά αποκλεισμένους από την οικονομική κρίση. Είχαμε κάποια συγκεκριμένα και σοβαρά συμπεράσματα, τα οποία υιοθετά, υιοθετήσαμε αργότερα. Όμω, τα πιο καλά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται στις προτεραιότητές μας, τα καταφέραμε να τα έχουμε τον Ιούνιο, τον Ιούνιο στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έλαβε χώρα πριν από μια εβδομάδα. Λοιπόν, το Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης έθεσε τρεις δείκτες οι οποίοι θα μπορέσουν να υπολογίσουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων κατά, καταπολέμησης της στόχιας. Λοιπόν, η ικανότητα να υπολογίσουμε όλες αυτές, όλους αυτούς τους δείκτες πραγματικά έγινε, θεωρήθηκε μια ιστορική πλέον συμφωνία και θέσαμε ως στόχο να καταφέρουμε να μειώσουμε ε, τη φτώχεια κατά 20 εκατομμύρια άτομα μέχρι το 2020. Εξού και το 2020. Γι' αυτό καταφέραμε ο αγώνας καταπολέμησης της φτώχειας να αποτελέσει μία από τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την... και βεβαίως ε, την έχουμε ονομάσει, όπως είπαμε, 2020, στρατηγική 2020. Όσον αφορά τον κοινωνικό αποκλεισμό και την καταπολέμηση τη φτώχεια, πρέπει επίσης να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση των γυναικών. Γιατί οι γυναίκες κινδυνεύουν πάρα πολύ από τη φτώχεια, περισσότερο από ότι οι άνδρες έχουν μικρότερου μισθού και βεβαίω πρέπει να δούμε το θέμα τους πολύ προσεκτικά, φροντίζουν τα παιδιά τους, εργάζονται ταυτόχρονα, η ζωή τους είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η Ισπανία ενδιαφέρεται επίσης η, στις πολιτικές έτσι, ενεργούς ένταξης και θέλει να δημιουργήσει μια στρατηγική γραμμή όλων των ε, κατευθυντηρίων γραμμών. Αυτά συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της διάσκεψης για την κοινωνική ένταξη που έλαβε χώρα τόνο στις Βρυξέλλες στις αρχές Μαΐου. Επίσης, θεωρούμε πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε την ανάγκη να φροντίσουμε τους άτομα που βιώνουν τη φτώχεια που είναι ε, ηλικιωμένα. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και αυτό. Και επίσης προσέξαμε πάρα πολύ τα θέματα που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες διότι και αυτοί επηρεάζονται πάρα πολύ από ε, το μη ευνοϊκό κλίμα των διαφόρων οικονομιών μας. Θα ολοκληρώσω αναφερόμενοι σε κάποιες σκέψεις που πιστεύω ότι μοιραζόμαστε όλοι. Η τρέχουσα κατάσταση της κρίσης και τα μέτρα τα οποία απαραίτητα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να την ξεπεράσουμε, δεν θα έπρεπε να δημιουργήσουν εμπόδια στην κατάσταση ευημερίας και στις κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές συνοχής. Δεν θα πρέπει ό,τι έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, τα τελευταία 20 χρόνια να μείνουν πίσω και πιστεύω ότι οι συμφωνίες στις οποίες θα καταλήξουμε αυτές τις μέρες θα οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου. Δεν θέλουμε μόνο να, είμαστε, να υποφελούμαστε από τις, πολιτικές, από τις κοινωνικές πολιτικές, αλλά θέλουμε να τις σχεδιάζουμε κιόλα. Θέλουμε να θέσουμε φιλόδοξους στόχους που θα μας βοηθήσουν και στο μέλλον. Ο κοινωνιολόγος Μπάουμαν από τη Γερμανία έλεγε ότι βασικά η τύχη μιας ε, κοινωνίας όπως και η δύναμη μιας ε, γέφυρας, η βάση μετριέται από τη δύναμη ε, πραγματικά που, που, που, που εμφανίζει. Και εγώ Συμφωνώ και θέλω να πω ότι πρέπει να ενισχύσουμε, να ενδυναμώσουμε αυτό το οποίο είναι η δική μας δύναμη ήδη υπάρχουσα. Έλεγα ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε να ενδυναμώνουμε την κοινωνία μας να ενδυναμώνουμε όλα τα στρώματα της κοινωνίας μας. Ο Ούλαφ Πάλμε έλεγε ότι η πολιτική, η προοδευτική πολιτική θέλει πάντα την αλλαγή, γιατί η αλλαγή υπόσχεται μια βελτίωση, τροφοδοτεί τη φαντασία και δίνει ενθάρρυνση σε όλα μας τα όνειρα, σε όλες τις αποστολές μας και τα οράματά μας. Και για μια προοδευτική πολιτική το μέλλον πάντα αποτελεί υπόσχεση μια ελπίδα. Το μέλλον δεν μπορεί να μας προκαλεί αβεβαιότητα και φόβο, αλλά να θεωρηθεί ένας, ε, μια περίοδος για ευκαιρίες. Και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου σε αυτήν την περίοδο κρίση που διανύουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, ο στόχο των κρατών μελών, των κυβερνήσεών μα, των κοινωνικών οργανώσεων, ο στόχο όλων λοιπόν θα πρέπει να ενδυναμώσει τις ικανότητες της κοινωνίας έτσι ώστε να κατακτούμε κάθε φορά περισσότερα ποσοστά ε, ελευθερίας, ισότητας και ευκαιρίες για όλους. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από το φόβο του μέλλοντος. Θα πρέπει να σταματήσουμε να φοβόμαστε, μην αρρωστήσουμε και χάσουμε τη δουλειά μας. Θα πρέπει να φοβόμαστε μην μείνουμε άνεργοι και δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Πρόκειται για κινδύνους της ζωής η ασθένεια, το γύρας, η ανεργία. Αυτά σήμερα είναι στόχοι για ένα κράτος ευημερίας. Είναι μια κατάκτηση των ευρωπαϊκών πολιτικών που δεν μπορούμε να χάσουμε. Η δημιουργία και η ενδυνάμωση αυτών των δικτύων κοινωνικής προστασίας αποτέλεσε προτεραιότητα στη δική μας πολιτική και γι' αυτό η κοινωνική πολιτική πρέπει να συνεχίσει να είναι μία από, τις, από, τα, από τα βασικά μας σημεία ταυτότητας ως Ευρωπαίοι. Ένα, μια ταυτότητα για όλους μας. Θέλω να σας συγχαρώ άλλη μια φορά και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες του διημέρου και ελπίζω ότι θα καταλήξετε σε πολύ καλές αποφάσεις και προτάσεις και ιδέες και συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε να συνεχίσουμε και εμείς ε, με θάρρος να συνεχίσουμε το έργο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία. Thank you very Ευχαριστούμε την κυρία Μαρτίνες για τις επισημάνεις της, δηλαδή ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις και να φροντίσουμε ότι όλοι όσοι βιώνουν τη φτώχεια θα πρέπει να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής. Κάτι που δεν είναι δεδομένο και θα πρέπει όπως καταλαβαίνετε όλοι εμείς να εργαστούμε για, την υλοποίηση αυτού, στόχο, αυτού του στόχου συγγνώμη, και τώρα με το κλείσιμο της Ισπανικής Προεδρίας ε, δεσμευτήκατε συγγνώμη, ότι ε, πρόκειται να συνεργαστείτε με, την, με τις επόμενες Προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση αυτών των στόχων. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Σάμουελ, ο οποίος είναι ε, αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης για την Απασχόληση και προσωπεί τον αρμόδιο επίτροπο. Γεια σας. Αγαπητοί φίλοι, πράγματι χαίρομαι ότι είμαι μαζί σας σήμερα εξ ονοματός ε, του Επιτρόπου κ. Άντορ και σε μια συνάντηση με τους ανθρώπους που βιώνουν τη φτώχεια. Ο κύριος Άντορ δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι μαζί σας σήμερα το πρωί, αλλά σας στέλνει τους θερμούς του χαιρετισμούς. Λοιπόν, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια πιστεύω ότι η συνάντηση έχει καταφέρει ουσιαστικά, ουσιαστικά αποτελέσματα, δηλαδή να διατηρήσει το θέμα της φτώχειας στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο όπως είπαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και εθνικό επίπεδο. Αυτές οι συνεδριάσεις παίζουν ένα σημαντικότατο ρόλο όσον αφορά την διαμόρφωση της στρατηγικής της, στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της καταπόλεμης της φτώχειας και η ενεργή συμμετοχή είναι καλό, καλοδεχούμενη. Και είναι πραγματικά απόδειξη το γεγονός ότι η κοινωνική πολιτική μπορεί να είναι αποτελεσματική εφόσον όσοι βιώνουν ε, τη φτώχεια συμμετέχουν στην διαμόρφωση αυτών των πολιτικών και πραγματικά Χαιρόμαστε για το γεγονός ότι είναι πλέον θεσμοθετημένη αυτή η συνάντηση. Έχει, έχουμε σημειώσει ουσιαστικούς πρόδους... και νομίζω ότι παρόλα αυτά απομένει πάρα πολύ ακόμα που θα πρέπει να γίνει. Η φετινή χρονιά είναι η Ευρωπαϊκή Χρονιά αφιερωμένη σε καταπολέμηση της φτώχειας και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει σαν στόχο να μειώσει την φτώχεια και να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και την έχει μετατρέψει αυτή την προτεραιότητα σαν κύρια προτεραιότητα. Τώρα, τι θέλουμε να πετύχουμε. Πιστεύω ότι ένας από τους πρώτους στόχους είναι να προωθήσουμε και να, μια, να προωθήσουμε μια καλύτερη κατανόηση ως προς τον κοινωνικό αποκλεισμό. Τι σημαίνει σε μια Ευρώπη που χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη ποικιλομορφία. Νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά να έχουμε τους ανθρώπους που βγαίνουν τη φτώχεια να είναι στο επίκεντρο αυτής της χρονιάς αφιερωμένης σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Εμείς ελπίζουμε ότι αυτή η χρονιά θα διαμορφώσει μια νέα δυναμική η οποία θα εξασφαλίσει και θα ενισχύσει την ενεργή συμμετοχή σε αυτόν τον αγώνα. Αυτό το ευρωπαϊκό έτος είναι πραγματικά αφιερωμένο στην ανάδειξη των δικαιωμάτων των ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια και αυτό το ευρωπαϊκό έτος καταπολεμά τα στερεότυπα και το, τους στιγματισμούς. Εμείς θα θέλαμε να στείλουμε ένα ισχυρό και σαφέστατο μήνυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι η καταπολέμηση της φτώχειας είναι μια κοινή ευθύνη και όλοι έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και θα πρέπει να ενισχύσουμε τον εφιστάμενο ε, την υφιστάμενη κοινωνική συμμαχία και πέραν από τους φορείς που ήδη παίζουν κάποιο ουσιαστικό ρόλο στην καταπολέμηση της κοινωνικής φτώχειας. Το ευρωπαϊκό έτος αποτελεί μια ευκαιρία για τους κοινωνικούς εταίρους, για τις επιχειρήσεις, για τα μέσα ενημέρωση, για την τοπική αυτοδιοίκηση, για, τις, ε, για, τους πολιτικούς, δηλαδή όλοι να θέσουν στο επίκεντρο το θέμα της φτώχειας και όχι μόνο το 2010 αλλά και έπειτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως καταλαβαίνετε έχει θέσει, και το έχω ξαναπεί σαν κύριο στόχο την εξάλληψη της φτώχειας και τουλάχιστον μείωση της φτώχειας και, την, ε, και της ενίσχυσης και, της, ε, και του κοινωνικού μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού. Η νέα στρατηγική της Ευρώπης 2020, σε συνεργασία επίσης και με τη συμφωνία που, στην οποία κατέληξαν οι Υπουργοί Απασχόλης, έχουν καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο στόχο για τη μείωση της φτώχειας. Και αυτός ο στόχος βασίζεται σε τρεις δείκτες. Πρώτον, η σχετική φτώχεια, η ηλική φτώχεια και επίσης η ενεργεία. Και ο στόχος είναι να αγγίξουμε τουλάχιστον 20 εκατομμύρια πολίτες, να τους βγάλουμε ε, από το κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. Όπως αναφέρθηκε από τους προλήσαντες η η ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν αυτόν τον στόχο στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής και πιστεύω ότι είναι μια συμφωνία ιστορικής σημασίας που ρίχνει τα θεμέλια για μια καινούρια πολιτική και επίσης ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα της κατάστασης, γιατί κακά τα ψέματα, η κατάσταση η οποία επικρατεί στα κράτη-μέλη ποικίλει. Εν πάση περιπτώσει, είναι μείζονη σημασία ότι η μάχη κατά της φτώχειας και κατά του κοινωνικού αποκλεισμού θα στηρίζεται σε φιλόδοξους στόχους και κυρίως επίσης και σε εθνικούς στόχους. Η μάχη κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και της εξάρτηση φτώχειας είναι αναπόσπαστο κομμάτι στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 με αποτελέσματα ορατά, χειροπιαστά για μια πιο δίκαιη Ευρώπη. Σε αυτή τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 η Κομισιόν έχει προτείνει καινούριες πρωτοβουλίες για μια πλατφόρμα ε, για την κοινωνική συνοχή και η θεμείωση της φτώχειας. Εμείς αυτή την πλατφόρμα θέλουμε να μετατραπεί σε ένα χειροπιαστό ε, δείγμα αλληλεγγύης το φθινόπωρο, η Κομισιόν θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα λειτουργεί και τι θα σκοπεύει αυτή η πλατφόρμα. Τώρα, θα πρέπει επίσης να προβληματιστούμε για το πώς οι φυστάμενες λειτουργίες και διαδικασίες για την κοινωνική προστασία θα υλοποιήσουν τους ε, προκαθορισμένους στόχους. Ο στόχος μας είναι ό,τι λειτουργεί να το κρατήσουμε και να το εμπλουτίσουμε με καινοτόμες νέες προσεγγίσεις η πλατφόρμα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού θα υποστηρίζει τις προσπάθειες και την πρόοδο που θα επιτελείται στο πλαίσιο της νέας, της νέας στρατηγικής 2020, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και επίσης να αναβαθμίσουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια. Επίσης αυτή η πλατφόρμα θα πρέπει να ενσωματώσει και άλλες πολιτικές όπως είναι το θέμα της υγείας, της εκπαίδευσης, της μετανάστευσης και επίσης τη λεγόμενη ε, ψηφιακή ατζέντα. Αγαπητοί φίλοι, ε, αυτή η επιτυχία της νέας στρατηγικής 2020 θα... Η επιτυχία αυτή εξαρτάται από την συμμετοχή όλων των φορέων και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό κατά πόσον θα υφίσταται συντονισμός ανάμεσα στους φορείς και επίσης στους ανθρώπους που βιώνουν τη φτώχεια. Εμείς συνεχώς θα προβαίνουμε στην διάχυση προτύπων ε, πετυχημένων παρεμβάσεων. Θα συνεχίσουμε με αυτή τη νέα δυναμική, ούτως ώστε να τροφοδοτείται αυτή η ελπίδα για τους ανθρώπους που βιώνουν τη φτώχεια είναι γεγονός ότι αυτό το ευρωπαϊκό έτος αφιερωμένο στην τη φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού έχει δημιουργήσει σε μια νέα δυναμική και έχουμε ακόμα ένα εξάμεινο. Θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε την κυρία Σάμβιλ, η οποία μας περιέγραψε τις αποφάσεις που πήραν η ε, και πρόεδρο των κυβερνήσεων σε σχέση με την καταπόλεμη της φτώχειας και το κοινωνικό αποκλεισμό στις επενδυμίες. Δηλαδή, ο στόχος είναι να βγάλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον 20 εκατομμύρια πολίτες, θα μίνιμουμ το ελπίζουμε και όχι σαν μάξιμουμ να ε, αποσυρθούν, απεμπλοκούν από την φτώχεια 20 εκατομμύρια πολίτες. Ευχαριστούμε για αυτή την υπενθύμηση και επίσης ακούσαμε για το νέο αυτό εργαλείο, την πλατφόρμα που θα διαμορφωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα προσπαθήσει να συγκεντρώσει όλες τις σωστές πολιτικές, τις βέλτιστες πρακτικές και να τις ενισχύσει με νέες ε, πολιτικές, με νέες προσεγγίσεις. Τώρα, θα ήθελα επίσης να παρουσιάσω τον Φερνάντο Λόπες, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας. Όπως καταλαβαίνετε είναι μια πάρα πολύ σημαντική επιτροπή με εκπροσώπους των κυβερνήσεων. Αλλά έχουμε λίγο παρεδέψει τα ονόματα της κυρίας Αγγέριος Φερνάντες, η οποία θα παρέμβει και στη δική μας συνεδρία, ο κ. Φερνάντες θα παρέμβει αύριο όμως στην Ολομέλεια. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Αντέλια Φερνάντες η οποία εκπροσωπεί την αντιπροσωπεία της ε, περσινής συμμετοχής ε, της Ισπανίας. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, αγαπητοί φίλοι από τις 27-28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήθελα να σας χαιρετήσω. Πράγματι, είναι σημαντικό να ακούγεται η φωνή των ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια και κυρίως να συμμετέχουν στις διαδικασίες για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων οι λεγόμενοι άνθρωποι που βιώνουν τη φτώχεια έχουν δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτές τις συνεδριάσεις. Νομίζω ότι πέραν από αυτήν την ε, θεσμική και θεμητή ε, συνάντηση και συμμετοχή σε αυτό το, σε αυτό το γεγονός. Θα ήθελα να πω ότι πέραν από αυτή τη συμμετοχή εγώ προσπαθώ σε καθημερινή βάση να εμπλουτίζω τις γνώσεις μου, να εμπλουτίζω την εμπειρία μου. ξέρετε, πιστεύω ότι αυτοί και που οι πιο εύποροι είναι πνευματικά φτωχοί. Δεν έχει σημασία αν φοράει κανείς ε, ακριβά ρούχα ή έχει πολυτελές αυτοκίνητο ε, ότι αυτός υλικά τέλο πάντων είναι πλούσιος. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι χάνουν την ουσία, χάνουν το, την ουσία της ζωής. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζήσει με ανθρώπους που έχουν άλλες προτεραιότητες, προτεραιότητες που σχετίζονται με το χρήμα, με το ακριβό αυτοκίνητο. Γιατί ταυτόχρονα υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν πώς θα πληρώσουν το νίκη, το, τα κοινόχρηστα, το ρεύμα, το, τα φαγητό τους κτλ. Δυστυχώς, ξέρετε, πολλές φορές είναι πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες που θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουν επιλογές ή να αγοράσουν τα φάρμακα ή να αγοράσουν ε, τρόφιμα. Κάποιοι θεωρούν ότι αυτό το πρόβλημα δεν τους αγγίζει. Αλλά δυστυχώς η οικονομική κρίση, η χρηματοπιστωτική κρίση ε, έρχεται και μας υπενθυμίζει ότι όλοι είμαστε ε, ευάλωτοι. Δεν υπάρχει κανείς το απειρόβλητο. Υπάρχουν σήμερα πολίτες που έχουν 50 λεπτά για να περάσουν ε, την ε, ημέρα. Και νομίζω ότι ο καθένας, όπως καταλαβαίνει, κανείς προβαίνει σε θυσίες και ίσως εδώ τουλάχιστον σε αυτό το χώρο υπάρχει μια αναγνώριση της συμμετοχής μας. Υπάρχει, μας ακούνε, μας εκτιμούνε και ανεξάρτητα δηλαδή από τις πολιτικές πεπιθήσεις μας, από τα πιστεύω μας. Όλοι έχουμε δικαίωμα για μια αξιοπρεπή ζωή και όταν μιλάμε για αξιοπρεπή ζωή δεν εννοούμε να, όλοι δικαίωμα να έχουμε στην επιβίωση, να έχουμε τουλάχιστον δικαίωματα σε συγκεκριμένα πράγματα, σε μια αξιοπρεπή ζωή, σε, σε, διακοπές, πρόσβαση στην κουλτούρα, να πηγαίνει κανείς στον κινηματογράφο, να αγοράζει ένα βιβλίο, δηλαδή να, να μην έχει αυτή την υποχρέωση να, να επιλέξει ανάμεσα σε δύο ε, συγκεκριμένα πράγματα. Και πιστεύω ότι οι διακοπές και η πρόσβαση στην κουλτούρα, στη μόρφωση, είναι βασικότατα δικαιώματα, ανεξάρτητα εάν κανείς είναι άρρωστος, άνεργος, συνταξιούχος. Σε μια, θα λέγα, ιδιώδη κοινωνία, εάν έχουμε δυνατότητα και εργαζόμαστε και μιλάμε πάντοτε για μια εξωπεπή δουλειά, μια δουλειά με ενδιαφέρουν και μια δουλειά που ανταποκρίνεται στις δεξιότητές μας, τότε πράγματι, τα πράγματα γίνονται κάπως πιο εύκολα. Αλλά αν δεν μπορούμε να εργαστούμε λόγω π.χ. ασθένεια, λόγω ανεργία, οικονομική ανεργία, λόγω συνταξιοδότηση, θα πρέπει το κράτο να παρεμβαίνει. Να μην υπάρχει μια υποχώρηση του, του επίπεδου ζωή μα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βρεθούν τις κατάλληλες απαντήσεις στην μεγάλη ποικιλομορφία των καταστάσεων. Δεν μπορούμε, ξέρετε, μόνο διάστατα να, να φεύγουμε πακέτα λύσεων που θα είναι κομμένα και ραμμένα στα ανάγκη όλων των ε, δικαιούχων. Η απασχόληση δεν είναι πάντοτε η, μαγική λύση για την κοινωνική επανένταξη. Αποτελεί όμως έναν σημαντικό σταθμό στην διαδικασία της Κοινωνική επανένταξη. Θα πρέπει μέσα αυτή, στο, στο πλαίσιο αυτής της συλλογική προσπάθειας όλοι μαζί να κινητοποιηθούμε και ξεκινώντα από αυτή τη συνεδρίαση. Έχουμε δυνατότητα να ανταλλάσσουμε εδώ τις εμπειρίες μας, έχουμε την ε, ευκαιρία να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας και ξέρουμε ότι όλα αυτά τα, προβλήματα είναι πολύπλοκα και δυστυχώς πολλές φορές οι πολιτικοί αγνοούν την ουσία των προβλημάτων μας. Θα πρέπει και εμείς να έχουμε το θάρρος να καταθέτουμε εδώ τις εμπειρίες μας. Και για να ολοκληρώσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους ε, εδώ συμμετέχουν σε αυτήν την συνάντηση, που είναι εδώ να ακούσουν τα προβλήματά μας και νομίζω ότι η συμμετοχή σας, η παρουσία σας εδώ αποτελεί ουσιαστική απόδειξη για το ενδιαφέρον που δείχνει στα προβλήματα μας και ευχαριστώ επίσης τους όλους υπεύθυνους για την όλη διοργάνωση που μου δώσαν την ευκαιρία εδώ να παρέμβω και ευχαριστώ εσάς, τους συμμετέχοντες και ε, τους παλαιότερους επίσης. Δεν πραγματικά με έχει αλλάξει άτομο αυτή η εμπειρία, δηλαδή το γεγονός ότι άκουσα εμπειρίες, άκουσα ανθρώπινες μαρτυρίες και πραγματικά εκ νέου εκ βάθους καρδιάς σας ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Mrs. Ευχαριστούμε για αυτή την ε, σημαντική ε, μαρτυρία και επίσης ότι θα πρέπει να έχουμε και τη, όχι μόνο το θάρρος και την δύναμη και το κουράγιο που ε, δείχνεται ε, ερχόμενοι εδώ στις Βρυξέλλες. Είναι, καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μια σκληρή έτσι, και δοκιμασία αλλά και προσπάθεια που κάνετε για να συμμετέχετε σε αυτήν την συνεδρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, αλλά θα ήθελα να καλέσω την κυρία Αντώνιο Καρπαρέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει εδώ στο πάνελ. η οποία θα μας αναφέρει ποιες είναι οι προτάσεις της Κομισιόν Επικεφαλής, η κυρία Καπαρέλη, της Γενικής Διεύθυνσης για την Κοινωνική Πολιτική και για την Κοινωνική Επανένταξη και θα μας ενημερώσει για τις προτάσεις της Κομισιόν, σχετικά και με τις προτάσεις που κάναμε εμείς πέρσι, στην περσινή μας συνάντηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για την, αυτή την όλη διαδικασία και τελικά μου έχετε αναθέσει μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή. Δηλαδή ακούσαμε εδώ ανθρώπινες μαρτυρίες. Εγώ θα κληθώ τώρα να εισέλθω λίγο σε κάποια πιο έτσι, λογιστική διάσταση. Δηλαδή, να προβώσουμε επί σε μια αξιολόγηση αυτής της ε, περίοδου, δηλαδή τα εννέα τελευταία χρόνια και ως συνήθω ξέρετε, δηλαδή, εξαρτάται το καθένας πόσο βλέπει το ποτήρι, μισό γεμάτο. Όσον αφορά τα θετικά, αυτό που θα πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε είναι μια δυναμική που έχει διαμορφωθεί, μια δυναμική, μια θέληση να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Αλλά από την άλλη άποψη, από την άλλη μάλλον, αν δούμε τα χειροπιαστά αποτελέσματα, εδώ υπάρχει μια απογοήτευση. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ευσυχάσουμε. Λοιπόν, θα σας ανατρέξουμε λίγο στο παρελθόν. Το 2008 η Γαλλική Προεδρία, η οποία είχε ενεργή έτσι, συμμετοχή όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, πήρε την προβουλία για την οργάνωση μιας συζήτησης οργανής τραπέζης για, την, για τον κοινωνικό αποκλεισμό σε υπουργικό επίπεδο και επίσης σε συνδυασμό με την συνάντησή σας. Δηλαδή πήγανε συμμετέχοντες το δικό σου εδώ, από το δικό σου meeting, πήγανε σε αυτήν την συνάντηση σε υπορικό επίπεδο. Και θυμάμαι ο κύριος Μάρτιν Χέρις από την οργάνωση Solidarity και τέλος πάντων πέραν από αυτή τη διαδικασία οι άνθρωποι που βιώνουν τη φτώχεια είπαν ότι ωραία τα λόγια αλλά δεν μπορούμε πλέον να περιμένουμε. Είναι καιρός για, για δράση, για, για και πραγματικά ήταν πάρα πολύ συγκινητικό γιατί υπάρχει αυτό το χάσμα ανάμεσα στις, στα λόγια και στις ε, πράξεις. Ίσως τώρα, ειδικά αυτή η απόφαση που αναφέρθηκε από τους προλαλήσαντες με τη νέα στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύω ότι πρόκειται για μια μεγάλη τομή σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας. Άρα σιγά σιγά γεφυρώνουμε το, χάσμα ανάμεσα στη φτώχεια, ανάμεσα στις λέξεις και στις ε, ε, πράξεις και διάβασα πρόσφατα το πόρισμα για την στρατηγική της Λισαβόνας και αναφέρεται ότι θα πρέπει να πάρουμε ουσιαστικά μέτρα για την εξάλληψη της φτώχειας καθορίζοντας στόχους, μετρήσιμους στόχους. Αυτό το πόρισμα της στρατηγικής της Λισαβόνας πριν από 10 χρόνια. Αυτό πραγματικά σας δείχνει το, το χάσμα που υφίσταται, που υπάρχει ανάμεσα στις προθέσεις, στις λέξεις και στις πράξεις και στις ε, ε, χειροπιαστές πρωτοβουλίες. Το πρώτο κατόρθωμα θα έλεγα της συνάντησής σας ε, είναι το εξής. Δίνει την φωνή στους ανθρώπους που βιώνουν τη φτώχεια και που εξέφρασαν αυτή την απογοήτευσή τους. Που είπαν ότι είναι, δεν μπορούμε πλέον να περιμένουμε. Και ξέρετε, και αυτό ήδη έχει ε, είχε ουσιαστικέ επιπτώσει στο, να δώσει, με το να δώσει μια νέα όθηση στους ε, πολιτικούς να πάρουν πιο γενναία μέτρα. Επίσης, να αναφέρουμε την ενίσχυση των δικτύων, όπως είναι το δικό σας δίκτυο, το EPN, το οποίο έχει συσφίξει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά επίσης και με άλλου ευρωπαϊκούς ε, φορείς. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι σημαντικό, γιατί ακούγεται πιο δυναμικά η φωνή σας όταν ε, ε, λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο αυτά τα κοινωνικά δίκτυα. Επίσης, τα προβλήματα και τα προβλήματα που συζητήθηκαν τα τελευταία χρόνια με την, στο πλαίσιο της ανοιχτής ε, διαδικασίες του αναφέρθηκαν ζητήματα όπως ο ελάχιστος μισθός, η ενεργή, η, η επανένταξη, η κοινωνική επανένταξη και επίσης η πρόσβαση σε υπηρεσίες, η κοινωνική επανένταξη, η πρόσβαση στην στέγη. Πραγματικά όλα αυτά τα ζητήματα πιστεύω χάρη στην δική σας ε, πρωτοβουλία και κυρίως χάρη στις συναντήσεις σας, όχι μόνο, αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε και άλλους φορείς, π.χ. φορείς που δραστηριοποιούνται στον αγώνα καταπολέμησης της ε, φτώχειας που, που τα παιδιά και τα λοιπά. Άρα με άλλα λόγια έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά απομένουν πολλά πολλά ε, θα πρέπει να γίνουν. Και μια ουσιαστική προσέγγιση έχει όμως αναπτυχθεί όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα και πιστεύω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας, η νέα συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας δίνει δυνατότητα να ε, έχουμε στη διάθεσή μας διευρυμένα εργαλεία και μέσα για την καταπολέμηση της φτώχειας θα ολοκληρώσω εδώ την παρέμβασή μου λέγοντας ότι φυσικά με την οικονομική κρίση μεγαλώνει η πρόκληση και η ανάγκη να παρέμβουμε αλλά τουλάχιστον να ξέρετε ότι η δική σας προσπάθεια δεν είναι άσκοπη και μπορούμε να βασιστούμε και στο δικό σας έργο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Καρπαρέλη. Πράγματι, σας ευχαριστώ για την ε, συμμετοχή σας και κυρίως για τις πρώτες απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επίτροπη που ήδη δόθηκαν. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ντανιέλ Ντύρξ, η οποία θα μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα κάποιων ερευνών που έχουν γίνει στον τομέα αυτό, δηλαδή της κοινωνικής πολιτικής. Good morning, uh, everybody. Καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ ότι βρίσκομαι εδώ και θα σας παρουσιάσω κάποια αποτελέσματα από τις μελέτες που έχουν γίνει σχετικά με τις συναντήσεις που λαμβάνουν χώρα εδώ κατόπιν πρωτοβουλία τη βελική κυβέρνηση. Η βελική κυβέρνηση, σα επαδημίζω, ήταν η πρώτη που πήρε την πρωτοβουλία για την οργάνωση αυτή τη συνεδρία. Και επίση, σε συνεργασία γίνανε αυτέ οι μελέτε με, το δίκτυο, με το δίκτυο καταπολέμησης της φτώχειας. Γιατί ο αντίκτυπος, μελέτης αντικ, για τον αντίκτυπο ε, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα που έχουν αυτές οι συναντήσεις, όπως καταλαβαίνετε είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν χρειάστηκαν να, να, να, να γίνουν πολλαπλές ε, διεργασίες για να προχωρήσουμε αυτή τη μελέτη. Δηλαδή όλοι όσοι συμμετείχαν τα εννέα τελευταία χρόνια σε αυτέ τι συναντήσει, να του βρούμε, να, κατα... να συγκεντρώσουμε κάποιο υλικό με τις καταθέσεις τους γιατί δεν ήταν εύκολο. Επαναλαμβάνω κάποιοι είχαν εξαφανιστεί. Βρήκαμε όμως ε, πολλούς ανθρώπους που συμμετείχαν στις ε, ε, συναντήσεις όλα, αυτό το, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη. Πρόκειται εδώ για προκαταρκτικά αποτελέσματα. Το τελικό πόρισμα με αναλυτικές έτσι, προσεγγίσεις παρουσιάσεις θα είναι κατά πάσα πιθανότητα έτοιμο το, περίπου στις αρχές Οκτωβρίου. Μία μελέτη λοιπόν για το αντίκτυπο αυτών των συνεδριάσεων ε, Ξεκινάμε με τους στόχους που θα πρέπει να εξυπηρετήσει αυτή η μελέτη και όπως καταλαβαίνετε έχουμε καταλήξει, μάλλον καταλήξαμε σε κάποιες ερωτήσεις, μπορείτε να τις δείτε εδώ στη, στις οθόνες. Η πρώτη ερώτηση είναι η εξής. Ο αντίκτυπος πάνω στο που βιώνουν τη φτώχεια. Δηλαδή αυτές οι συναντήσεις κατά πόσον έχουν βοηθήσει στην καθημερινότητα τους ανθρώπους. Δεύτερη ερώτηση, ο αντίκτυπος πάνω σε άλλους ε, φορείς, σε, ακόμα και σε θε, θεσμούς, σε ιδρύματα. Προλαλήσαντες εδώ παρεμβαίνοντας, είπαν ότι πρόκειται εδώ για μια συλλογική μάχη η οποία θα πρέπει να ενώσει, να συγκεντρώσει όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Άρα όχι μόνο οι μη κοινωνικές οργανώσεις αλλά και οι θεσμοί. Επίσης, επιπτώσεις, ε, τρίτη ερώτηση, θα θέλαμε να μάθουμε ποια είναι τα αποτέλεσματα σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτών των συναντήσεων. Και τελευταία ερώτηση, σε σχέση με τις τρει τρεις πρώτες ερωτήσεις, η τέταρτη ερώτηση λοιπόν ε, εστιάζει πάνω στην αξιολόγηση της συμμετοχής, της δικής σας συμμετοχής σε αυτές τις συναντήσεις. Έχουμε λοιπόν μάλλον καταλήξαμε σε διαφορετικές μεθοδολικές προσεγγίσεις για να βρεθούν οι απαντήσεις και κυρίως να αγγίξουμε τους συμμετέχοντες και όσοι μπορούν να μας βοηθήσουν στο να, στο να, στην, να καλύψουμε αυτές τις ερωτήσεις. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση, ή μάλλον το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου, το οποίο η αναπτυξη του αριθματολογιου ίντερνετ Προχωρήσαμε, προσπαθήσαμε δηλαδή να συγκεντρώσουμε στοιχεία, email και καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο να αγγίξουμε περίπου 300 άτομα και μέχρι σήμερα 79 απάντησαν σε ερωτήσεις του εκμετολογίου μου. Ποιοι απάντησαν σε αυτές τις ερωτήσεις. Όπως καταλαβαίνετε σε μια πρώτη φάση κυρίως ήταν θεσμικοί παράγοντες, μη κυβερνικέ οργανώσεις, άνθρωποι που βιώνουν τη φτώχεια, οι υπεύθυνοι εδώ οι διοργανωτές της συνάντησης και ακαδημαϊκούς. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, ε, είναι πολύ δύσκολο να περιοριστεί κανείς όταν θέλει να απαντήσει σε μια, μια τέτοια ερώτηση. Ε, επειδή συνήθως αυτές οι απαντήσεις είναι διαμορφωμένες με κλειστό τρόπο. Δεν μπορεί κανείς να επιφέρει αποχρώσεις, να δώσει κάποιε λεπτομέρειες. Γι' αυτό το λόγο μετά φροντίσαμε να γίνουν κάποιες ε, συνεντεύξεις με τους ε, ε, συμμετέχοντες σε αυτήν την έρευνα. Και είχαμε ένα δείγμα από μη κυβερνικέ οργανώσει, από θεσμικούς παράγοντες και τα λοιπά, να απαντήσουν σε αυτές τις συνεντεύξεις. Και επίσης είχαμε εγώ σε συνεργασία με τον Νίκολας Βανχέλ, δύο ερευνητές πήγαμε, μας καλέσανε μάλλον σε πέντε χώρες να επισκεφθούμε ε, αυτές τις χώρες και να, να έρθουμε σε επαφή με υπεύθυνου και να συγκεντρώσουμε και άλλο υλικό σχετικά με αυτά τα θέματα. Και πέραν από αυτή την έρευνα που έγινε στο διαδίκτυο, μας έδωσε αυτή η ευκαιρία να μιλήσουμε, να έρθουμε σε επαφή με τους ανθρώπους, ακόμα πιο πλούσιο υλικό που συμπληρώνει το υλικό και το αποτέλεσμα που προέκυψε από την έρευνα στο ίντερνετ. Λοιπόν, τα πρώτα αποτελέσματα σας είπα είναι προκαταρκτικά και για η πρώτη ερώτηση είναι η εξή. Κατά πόσον αυτέ οι συναντήσει έχουν οδηγήσει με καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που βιώνουν τη φτώχεια. Ε, λοιπόν, τα πρώτα αποτελέσματα λένε ότι αναδεικνύουν το εξή. Το 79% των ε, ανθρώπων που απάντησαν απάντησαν μάλλον με θετικό τρόπο. Δηλαδή ότι καταλαβαίνουν καλύτερα τα προβλήματα των ανθρώπων που βιώνουν την φτώχεια. Αυτό είναι σημαντικό εφόσον θέλεις να διαμορφώσεις κατάλληλε πολιτικές. Δεύτερη ερώτηση, κατά πόσον έχετε μάθει, έχετε πάρει περισσότερες γνώσει ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα καταπολεμήσετε τη φτώχεια. Και το 80% των πολιτικών απαντά ότι ναι, πράγματι έμαθε πολλά πράγματα στο πλαίσιο για το, για σκοπό της καταπολέμησης της φτώχειας και κυρίως ότι από αυτές τις συναντήσεις έχουν αλλάξει τον τρόπο τον οποίο προωθούν τις πολιτικές τους. Και αυτό έρχεται σαν τη διαστολή με, τους, ε, με τις απαντήσεις από τους άμεσα ενδιαφερόμενους οι άνθρωποι που βιώνουν φτώχεια λέει εγώ δεν έμαθα περισσότερα πράγματα από τη συμμετοχή μου σε αυτές τις συναντώσεις όσον αφορά την, τα προβλήματα της φτώχειας. περίπου είναι στο 56% αυτών των ανθρώπων. Ε, επίσης αναγνωρίζει ότι άλλαξε και την καθημερινότητα ε, αυτή η συνάντηση, η συμμετοχή σε αυτές τις συνεδρίες. Λοιπόν, το επόμενο θέμα έχει να κάνει με το πώς επωφελήθηκαν από αυτή τη συνάντηση. Ειδικά από την Λιθουανία είχαμε μια πολύ δυναμική συμμετοχή και ειδικά στην ερώτηση κατά πόσον αυτή η συνάντηση σας βοήθησε προσωπικά, πρώτη ερώτηση και δεύτερη ερώτηση, κατά πόσον σας έδωσε δυνατότητα να αναπτύξετε σχέση αλληλεγγύης με τους υπόλοιπους άνθρωπους που βιώνουν τη φτώχεια. Εδώ έχουμε φωτογραφίες από την Πολωνία και 87% ε, ε, των ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια θεωρούν ότι αυτές οι συναντήσεις έχουν βελτιώσει την ε, προσωπική τους ανεξέλιξη. Και ειδικά το κομμάτι της αυτοπεποίθησης, της αποκατάστασης της αυτοπεποίθησης των συμμετοχόντων. Δηλαδή θεωρούν ότι ε, εφόσον φεύγουν από αυτή τη συνάντηση έχουν, ε, αποκτούν μεγαλύτερο έτσι, θάρρος, κουράγιο για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους και τέλος πάντων με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση θα ε, αντιμετωπίσουν πλέον τα προβλήματά τους μια άλλη ε, πτυχή αυτής της προσωπικής ανεξέλιξης που ανα... στην οποία αναφερόμαστε είναι το συναισθημα... κομμάτι. Δηλαδή υπάρχει έτσι μια συναστηματικη εκπλήρωση με την έννοια ότι πλέον οι άνθρωποι που βιώνουν τη φτώχεια δεν θεωρούν ότι είναι απομονωμένοι μετά την συμμετοχή τους σε αυτή τη συνάντηση και επίσης το δικαίωμα για σεβασμό και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή το γεγονό ότι ακούγεται η φωνή του. Τώρα, επόμενη ερώτηση είναι η ελεγγύη. Το 50% των ε, ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια θεωρεί ότι συμφωνεί με αυτήν την ε, διατύπωση. Με άλλα λόγια, θεωρούν ότι πρόκειται για μια ε, έτσι διαφέρουσα εμπειρία να μαθαίνεις το πώς οι άνθρωποι από άλλες χώρες βιώνουν τη φτώχεια. Πρώτον και το να μαθαίνω ότι όχι μόνο στη χώρα μου υπάρχουν προβλήματα με κοινωνικό αποκλεισμό και με φτώχεια, αλλά υπάρχουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες προβλήματα που συνδέονται με τον κοινωνικό αποκλεισμό. Και επίσης το πώς προσπαθούν οι, οι, άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Δηλαδή υπάρχει μια ανταλλαγή απόψεων και, και κατά πόσον επίσης αναβαθμίζεται η σχέση εμπιστοσύνη με τους ε, πολιτικούς. Επίσης, προσπαθήσαμε να δούμε ποιος είναι, πώς διαμορφώνεται ο αντίκτυπος τους ε, θεσμικούς φορείς και στους πολιτικούς και περίπου το 40% θεωρεί εδώ των συμμετεχόντων ότι αλλάζουν ε, οι πολιτικές των θεσμών. Οι μη κυβερνικέ οργανώσει πράγματι το περίπου 50% των μη κυβερνικών οργανώσεων θεωρούν ότι μας έχει δώσει μια νέα ακόμα πιο δυναμική όθηση, το να δηλαδή η συμμετοχή μας σε αυτές τις συναντήσεις, μας έχει δώσει μια νέα όθηση για να καταπολέμησουμε την φτώχεια. Και επόμενες ε, ερωτήσεις ή μάλλον διατυπώσεις κόκκινο χρώμα είναι να, να αναφέρεται στην ανάγκη ότι χρειάζεται μια δημόσια συζήτηση. Μια δημόσια συζήτηση που θα εξασφαλίσει ότι η φτώχεια είναι στο επίκεντρο της ατζέντα της ε, χώρας μας. Τώρα, πράσινο χρώμα, κάποιες πιο θετικές έτσι, παρατηρήσεις. Δηλαδή από αυτή την ε, πλέον θεσμοθετημένη συνάντηση προέκυψαν νέες οργανώσεις, ενώσεις που διαμορφώθηκαν, σχηματίστηκαν πάντοτε με στόχο της καταπολής πτώχειας Και επίσης από αυτές τις συναντήσεις προέκυψαν νέες συνέργειες, νέες ε, συνεργασίες και κυρίως βελτιώθηκε η, και ποσοτικά και ποιοτικά η ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Impact on the policies. Αντίκτυπος στις πολιτικές. Σχεδόν το 60% των υπεύθυνων χάραξης πολιτικών πιστεύουν ότι υπάρχει πραγματικά αντίκτυπο στις πολιτικές, αλλά το 78% των ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια δεν το πιστεύουν, δεν θεωρούν ότι επηρεάζονται οι πολιτικές. Συνεπώς, πρέπει να βρούμε ποια είναι η διαφορά και πώς μπορεί αυτή η διαφορά να εξηγηθεί. Ενδεχομένως να υπάρχει αντίκτυπο στις πολιτικές, αλλά τελικά να μην αγγίζει αυτός ο αντίκτυπος τους ίδιους τους ανθρώπους που βιώνουν τη φτώχεια. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι αυτές οι συνεδριάσεις βοηθούν και ενθαρρύνουν την ε, εκπόνηση μέτρων. Κάποια παραδείγματα του αντίκτυπου των πολιτικών που είχαμε στην έρευνά μας. Πρώτον, οι πολιτικοί έμαθαν τι κρύβεται πίσω από τα νούμερα. Συγκεκριμένα ότι η φτώχεια έχει να κάνει με την πραγματική ζωή. Τι σημαίνει δηλαδή να ζει κανείς στη φτώχεια. Ε, ποιες είναι οι εμπειρίες, ε, γιατί αγωνίζονται καθημερινά οι άνθρωποι. Ένα από τα αποτελέσματα λοιπόν είναι αυτό. Επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι η δημιουργία μέσα σε αυτές τις ε, συνεδριάσεις το θέμα της φτώχειας μπήκε στην ατζέντα και οι πολιτικοί άρχισαν και συνέχισαν να μιλούν για το θέμα ε, της φτώχειας και της καταπολέμησής της. Πιο συγκεκριμένα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε κάποια αποτελέσματα, π.χ. τη στρατηγική της φτώχειας 2020, ή κάποιε άλλε συστάσεις για την κοινωνική ένταξη, πράγμα που είχε συζητηθεί εδώ πέρα στη συνεδριάσει και μετά συνεχίστηκε το επίπεδο συζητήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. το Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Στόχιας το 2010. Επίσης έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι υπάρχει σχέση μεταξύ αυτών των συνεδριάσεων ε, και του ειδικού ε, της ε, ανοιχτής μεθόδου διαπραγματεύσεων. Συζήτηση επίσης για την ενεργειακή φτώχεια, ένα άλλο θέμα που τέθηκε εδώ πριν από μερικά χρόνια. Σε εθνικό επίπεδο χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο, περισσότερα δεδομένα που θα συλλέξουμε τους επόμενους μήνες για να δούμε μέσα από μελέτες περιπτώσεων τον αντίκτυπο σε εθνικό επίπεδο. Τώρα όμως μπορούμε να πούμε π.χ. ότι στην Ιταλία η συνάντηση των ανθρώπων που βιώνουν την ε, φτώχεια χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα προκειμένου να διοργανωθούν εθνικές πρακτικές και συνεδριάσεις. Οι εθνικές ε, συναντήσεις λοιπόν με τη σειρά τους επίσης οδήγησαν σε μια πολύ καλή προετοιμασία για αυτήν εδώ την ευρωπαϊκή συνάντηση. Και βεβαίως Κάποια άλλα παραδείγματα ετέθησαν σχετικά με την κατάσταση των ε, Ρώμα στις διάφορες χώρες, στα προβλήματα της ενέργειας. Τελευταίο σημείο έχει να κάνει με τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις. Τα αποτελέσματα είναι γενικώ πολύ θετικά. Πάρα πολλές ερωτήσεις έχουν τεθεί ε, και μάλιστα ψήν 75% είναι το αποτέλεσμα και βλέπετε εδώ η βελγική αντιπροσωπεία είναι πολύ ευτυχισμένη στη φωτογραφία. Δεν συμφωνούν. Επίσης, όσον αφορά τη συμμετοχή, το θετικό είναι ότι οι άνθρωποι αναγνωρίζουν ότι πραγματικά έχουν κίνητρα ε, υπάρχει μια καλή προετοιμασία. Δεν στρεσάρονται πάρα πολύ, δεν έχουν προβλήματα συμμετοχής, ούτε γλωσσικά, ούτε τίποτα άλλο. Και γενικώ όσον αφορά τα αρνητικά, είπαμε ότι μερικέ φορέ ο κόσμο είχε πολύ ψηλέ προσδοκίε από τη συνάντηση και έτοιμο για περισσότερη συμμετοχή από εθνικούς πολιτικούς ηθήνοντες. Παρουσία εδώ αυτών των ανθρώπων έτσι ώστε να εμβαθύνουμε πιο πολύ στα θέματα. Και για να ολοκληρώσω θέλω να σας δείξω αυτή την κοινική έτσι, εικόνα. Σε αντίθεση όμως με αυτό το κοινικό σκηνικό που βλέπετε, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα καλό μέλλον για τη, για τη συνέχιση αυτών των ευρωπαϊκών συνεδριάσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που μας τονίσατε όλα αυτά τα θέματα και που αρχίσατε να δίνετε κάποιες απαντήσεις. Γιατί το ερώτημα που τίθεται πολύ συχνά είναι τι μας αποφέρει μια τέτοια ευρωπαϊκή συνάντηση. Και νομίζω ότι ήδη έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι βλέπουμε ότι οι αντιλήψει είναι πολύ διαφορετικές μερικές φορέ μεταξύ των ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια και μεταξύ των ε, υπεύθυνων χάραξη πολιτικών. Βλέπουμε το υψηλό ποσοστό συμμετοχής και νομίζω ότι είναι ενθαρρυντικό το να γνωρίζουμε ότι πραγματικά και για τους πολιτικούς ευθύνοντες ε, υπάρχουν αποτελέσματα μέσα από αυτές τις συναντήσεις. Και αυτό είναι και πιο σημαντικό γιατί γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ. Ερχόμαστε από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, θέλουμε να βελτιώσουμε τις πολιτικές. Και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο μας το αποδεικνύει η συγκεκριμένη μελέτη. Λοιπόν, έχουμε ξεφύγει λιγάκι από το χρόνο μας, όμως δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία να σας δώσω το λόγο και σε εσά και να ακούσω ενδεχομένως κάποιες αντιδράσεις που μπορεί να έχετε βάσει ε, των παρεμβάσεων των ε, εισηγητών μας. Ε, δεν θα μακρηγορήσουμε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που θέλει το λόγο. Βλέπω εδώ ένα χέρι να σηκώνεται. Ωραία, έχω ήδη τρεις λοιπόν παρεμβάσεις, τέσσερις. Για την ώρα στις τέσσερις παρεμβάσεις θα παραμείνουμε. Καταρχάς από αυτή την πλευρά παρακαλώ. Μάλιστα, θα ήθελα να κάνω μία πρόταση. Οι ευρωπαϊκές συναντήσεις δεν θα πρέπει να ε, λαμβάνονται υπόψη με ξεχωριστό τρόπο. Θα πρέπει να παραμένουν στην, Ευρω... στην ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χρειάζεται μια νέα στρατηγική, ένα νέο στρατηγικό ε, σχέδιο για το 2020. Γι' αυτό το σκοπό θα πρέπει να δημιουργηθεί η πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας με μια άμεση ενσωμάτωση και ένταξη των ανθρώπων των ίδιων που βιώνουν τη φτώχεια. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ε, καλό θα είναι να, να λέτε τη γλώσσα στην οποία θα μιλήσετε, θα εκφραστείτε και να συστήνεστε. Βεβαίως ήταν η Μαρή Λουίς Δεκχόκ από τη Βελγική Αντιπροσωπεία, η οποία πήρε το λόγο. Επειδή και ο ίδιος είμαι Βέλγος, τη γνώριζω καλά, γι' αυτό και μπόρεσα να, στη, να σας τη συστήσω. Παρακαλώ, η γερμανική αντιπροσωπεία έχει το λόγο. Είμαι ο Γιάννης Στογάιντερ από, την ε, από τη γερμανική αντιπροσωπεία. Λοιπόν, σήμερα το πρωί ακούσαμε πάρα πολλές παρεμβάσεις. Συμπέρασμα. Η πρόκειται για την ίδια διαδικασία με πέρσι. Από την άποψη των πολιτικών ακούμε ότι θέλετε να υλοποιήσετε τις ιδέες μας, αλλά δεν κάνετε τίποτα γι' αυτό. Π.χ. η κρίση είχε πολύ σοβαρές συνέπειες. Οι κερδοσκόποι, οι πλούσιοι, οι τράπεζες, αυτοί έλεγαν δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Σήμερα αυτές οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σκοπεύουν να εφαρμόσουν νομοθεσίες μέσα από τις οποίες εμείς θα πληρώσουμε την ύφη, φτωχή. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν είναι οι, εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια φορά σοβαρά να λάβουν υπόψη τα συμφέροντά μας και όχι μόνο να έρχονται εδώ να μας ακούνε και να λαμβάνουν μετά υπόψη μόνο τα οικονομικά τους συμφέροντα. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, ο κύριος... Ναι. Έχετε το λόγο. Πέδρο ε, Γκονσάλβος, ε, Από την Πορτογαλία. Καταρχάς, Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παρόντες εδώ, όλους αυτούς που βιώνουν τη φτώχεια, γιατί πραγματικά είναι οι πρωταγωνιστές της Ευρωπαϊκής Συνεδρίασης. Χωρίς αυτούς τους ανθρώπους δεν θα βρισκόμασταν εδώ. Ε, εδώ και αρκετό καιρό συζητάμε δεν ξέρω για πόση ώρα δηλαδή, αλλά για αρκετή ώρα μιλάμε για στατιστικά στοιχεία, για στρατηγικές, για μελέτες, Μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια. Πολλοί άνθρωποι δεν είχαν την ευκαιρία ούτε καν να, φάνε σήμερα. Δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι χειρότερα από μας. Πρέπει να ευθυγραμμίζουμε τα στατιστικά στοιχεία, τις ε, θεωρίες με την πρακτική. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι απελπισμένοι, που βιώνουν πολύ έντονα τη φτώχεια, βιώνουν τη μόνιμη αγωνία και όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι αντικείμενα. Ε, δεν πρέπει να πάντα να αγοράζουμε ε, εξοπλισμούς, ε, όπλα, να φτιάχνουμε αεροδρόμια. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά χρειάζεται να φροντίσουμε και τους ανθρώπους. Εδώ δεν είμαστε υλικό, δεν είμαστε αντικείμενα, μιλάμε για ανθρώπους. Να το καταλάβουμε αυτό και εδώ λοιπόν σας προκαλώ ανοιχτά να δημιουργήσουμε μία χάρτα των δικαιωμάτων των ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια. Δικαιώματα και υποχρεώσεις, δεν λέω. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε, όπως και εσείς το κάνατε, και ο Γιάννης του άλλους πριν από εσά, από την γερμανική αντιπροσωπεία το έκανε, ότι έχει σημασία να εξετάσουμε και άλλου τομείς, όχι μόνο τα κοινωνικά θέματα. Ε, όπως αναφέρθηκε λοιπόν, να δούμε και τον προπολογισμό. Και ο προπολογισμό είναι σημαντικό, δηλαδή πού πάνε τα χρήματα. Πηγαίνω πίσω λοιπόν στην αίθουσα στο πίσω μέρος, παρακαλώ. Γεια σας, είμαι από την Μάλτα και θα μιλήσω ε, μαλτέζικα. Πολύ συχνά μιλάμε για την εξάλληψη της φτώχειας. Πολύ καλή ιδέα, αλλά πρέπει να προσέξουμε. Ενδεχομένως να δώσουμε την εντύπωση ότι κάποια μέρα πρέπει να σταματήσουμε να καταπολεμούμε. Όχι, η μάχη μας θα πρέπει να είναι διαρκής, γιατί οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες αλλάζουν διαρκώς. Άρα η ιδέα ότι ίσως κάποια μέρα να, χρεια... να μπορέσουμε να σταματήσουμε να καταπολεμούμε τη φτώχεια δεν είναι ρεαλιστικό πράγμα. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο άκουσα. Εντυπωσιάστηκα γιατί άκουσα ότι υπάρχουν διαφορές ε, μεταξύ των τομέων της κοινωνικής και της οικονομικής πολιτικής και ότι οι στρατηγικές και οι πολιτικές πολλές φορές δεν ταιριάζουν. Αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερος. Και ο λόγος είναι ότι η πολιτική με όλες τις προτάσεις πρέπει να είναι ολιστική. Με άλλα λόγια. Πρέπει να θυμόμαστε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με πραγματικούς ανθρώπους, με πραγματικές ζωές. Πρέπει να έχουμε επίση κατά νου και την ευρύτερη διάσταση, την πολιτική και την οικονομική. Συνεπώς, ναι, πρέπει να επιμείνουμε ως προς τη σημασία του ελάχιστου εισοδήματο. Ναι, πρέπει να δούμε ότι και η βιομηχανία θα πρέπει να κινηθεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους, όχι για νούμερα και στατιστικά στοιχεία. Είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να δουλέψουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι δεν θα έχουμε το χρόνο να δώσουμε το λόγο σε όλους όσοι σήκωσαν το χέρι. Αλλά κατά τη διάρκεια των ομάδων εργασίας θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις και όλοι λίγο πολύ θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε το λόγο. Η κυρία Φεντερίκο έχει τελευταία το λόγο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω ισπανικά, είμαι από την Ισπανία εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση καταρχάς. Γιατί αυτοί, αυτές οι συναντήσεις δεν καταλήγουν εκεί που θέλουμε. Εγώ δηλαδή δεν ήξερα καν ότι υπήρχαν αυτές οι ευρωπαϊκές συναντήσεις μέχρι φέτος. Γιατί δηλαδή ε, δεν δε, γίνεται γνωστό τι αυτή η Ευρωπαϊκή Συνάντηση. Και να πω το εξή. Η φτώχεια, όχι μόνο η οικονομική φτώχεια, ε, σημαίνει και μη πρόσβαση στον πολιτισμό. Μη πρόσβαση στην αποσχόληση. Εμένα κανείς δεν θα με προσλάβει επειδή είμαι σαν απειρικό καροτσάκι. Εντάξει, υπάρχει οικονομική φτώχεια αλλά υπάρχουν και άλλα είδη φτώχειας. Και εγώ είμαι φτωχή, έχω να φάω, αλλά δεν έχω πρόσβαση σε μια σειρά πραγμάτων που προσφέρει κανονικά η κοινωνία. Οπότε, πρώτον, ερώτηση, γιατί δεν ενημερωνόμαστε για τέτοιου είδους ευρωπαϊκές συναντήσεις και δεύτερον, να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει μόνο οικονομική φτώχεια. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Να θυμόμαστε ότι δεν είναι μόνο τα χρήματα, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη φτώχεια. Τώρα, η κυρία Φιγκουρέλο έχει το λόγο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω όλους τους παρόντες εδώ στη συνεδρίασή μας και παρά τις επικρίσεις που ακούστηκαν θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είστε όλοι σημαντικοί και έχει σημασία να έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάσσουμε εμπειρίες, να ακούμε τις διάφορες πτυχές του προβλήματος. Συμφωνώ όμως, πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω. Δεν φτάνει αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι που βιώνουν τη φτώχεια είναι κουρασμένοι. Κουρασμένοι από λόγια, λόγια χωρίς καμία δράση. Θέλουν δράσεις, μέτρα πρακτικά, συγκεκριμένα πράγματα. Και πιστεύω ότι εδώ βρίσκεται το μεγάλο διακύβευμα, μεγάλη πρόκληση για τους πολιτικούς ηθήνοντες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το 2010 είναι η Ευρωπαϊκή Χρονιά για την καταπολέμηση της στόχιας από τη στιγμή που στη συνέχεια αποφασίζουμε να υλοποιήσουμε προγράμματα λιτότητας προκειμένου να σεβαστούμε το σύμφωνο σταθερότητας και να μειώσουμε τον προπολογισμό. Όταν μειώνουμε τον προπολογισμό, πραγματοποιούμε μειώσεις στον δημόσιο τομέα, στις δημόσιες υπηρεσίες, ε, στην κοινωνική βοήθεια. Άρα τι κάνουμε, παρατείνουμε το όριο συνταξιοδότησης, μειώνουμε τον ελάχιστο μισθό, αυξάνουμε τη φορολογία του εισοδήματο. Αυτό δεν γίνεται, είναι αδύνατον. Και όμως ε, ε, εδώ βρισκόμαστε. Δηλαδή ε, έχουμε το έτος καταπολέμησης της στόχιας και ταυτόχρονα οι οικονομικές πολιτικές επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση και το βάρος του σώμου των ανθρώπων γίνεται ανυπόφορο. Αυτό αποτελεί πραγματικό σκάνδαλο. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να εκφραστούμε. Να μιλάτε. Να μιλάτε για, για τους πολιτικούς, αλλά μην τους βάζετε όλους στο ίδιο καλάθι. Υπάρχουν πολιτικοί που είναι με, την, με, με με το μέρος σας και πραγματικά προσπαθούν ε, να, να σας βοηθήσουν. Η κυρία από την ε, Κοινωνική Επιτροπή είπε ότι χθε ε, ψηφίσαμε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και α, Απασχόλησης μία έκθεση η οποία τονίζει αυτά τα προβλήματα και η οποία κρούει τον κόδωνα κινδύνου. Δυστυχώς παρά το γεγονός ότι εγώ είμαι μία από τις βασικές εισηγήτριες και παρόλο που έχω δικαίωμα ψήφου, η πλειοψηφία αποφασίζει. Παρά το ρόλο μου όμως, η έκθεση δεν με ικανοποιεί πλήρως και θα σας θέσω μια νέα πρόκληση. Η έκθεση αυτή θα, θα ψηφιστεί τον Οκτώβριο στην Ολομέλεια. Μια νέα συζήτηση θα λάβει χώρα στην Ολομέλεια και μέχρι τότε έχετε τη δυνατότητα να προτείνετε αλλαγές προκειμένου να βελτιωθεί αυτή η έκθεση και να πούμε στο, στην Κομισιόν και στο ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ήρθε η ώρα για δράσεις και όχι για λόγια. Πρέπει να εγγυηθούμε υπηρεσίες για όλες και όλους, πρέπει να εγγυηθούμε ελάχιστο εισόδημα για όλες και όλους που μας επιτρέπει να ζούμε αξιοπρεπώς και έχουμε ξαναμιλήσει στα πλαίσια αυτών των συνεδριάσεων δεν πρόκειται απλώς για χρήματα έτσι ώστε να έχουμε ένα πιάτο φαΐ, αλλά να μπορούμε να εξασφαλίζουμε και την παιδεία μας, μια αξιοπρεπή στέγαση, πρόσβαση στα πολιτιστικά δρόμενα κτλ. Οι φτωχοί έχουν και αυτοί δικαίωμα στην κουλτούρα, στον πολιτισμό. Είναι απαραίτητο λοιπόν το ελάχιστο εισόδημα να προσαρμοστεί και να αποτελέσει κανόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται ευρωπαϊκός νόμος για να τα καταφέρουμε. Χθε δεν καταφέραμε να το συμπεριλάβουμε αυτό στην έκθεση, όμως είμαι βέβαιο ότι με τη δική σας βοήθεια θα τα καταφέρουμε μέχρι τον Οκτώβριο. Όλοι και όλες πρέπει να δουλέψουμε σκληρά προκειμένου να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Όμως, αυτό θα αποτελέσει το πρώτο βήμα μόνο. Μετά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η έκθεση αυτή ε, γίνεται και πρακτική και καλύπτει όλους τους ανθρώπους που βιώνουν τη φτώχεια. Πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι φτωχοί να μην είναι πλέον φτωχοί εργαζόμενοι. Να υπάρχει εγγύηση μισθών, αξιοπρεπών ε, θέσεων εργασίας, με αξιοπρεπείς συνθήκες και μισθούς. Ε, οι συνταξιούχοι που ζουν στη, στη φτώχεια και αυτοί έχουν δικαίωμα να έχουν επιδόματα αξιοπρεπή επιδόματα. Θα πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσουμε τις πολιτικές της Κομισιόν και του Συμβουλίου και αυτή είναι η πρόκληση που σας καταθέτω και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε ακόμη περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Ήθελα απλώς να σας εκφράσω την υποστήριξή μου και τη βοήθειά μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Φιγκιουρέιντο. Ακριβώς μας εξηγήσατε πόσο σημαντική είναι η συνεργασία όλων μας και δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο, πρέπει να κλείσω τη συζήτηση της Ολομέλειας. Θα συνεχίσουμε όμως το διάλογό μας στις επόμενες ε, συνεδριάσεις, μετά από το διάλειμμα. Πριν πάμε όμως αυτό, θέλω να δώσω το λόγο στην Μισελίν Ζεγοντάλ για κάποιες πρακτικές ανακοινώσεις και Ακούσατε πολλά τους τελευταίες μήνες από την Μισλίν και γι' αυτό θέλω να την ευχαριστήσω για όλη τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε προκειμένου να διοργανώσει τη συνεδρία. Ευχαριστούμε Μισλίν. Alors, quelques... Λοιπόν, κάποιες πρακτικές πληροφορίες. Λοιπόν, για να βρείτε την ομάδα εργασίας σας στο τέλος του διαλύματος του καφέ. Πρέπει να ακολουθήσετε τη φωτογραφία του κοριτσιού που κοιτάζει ατενίζει το μέλλον. Θα δυσκολευτείτε λιγάκι, αλλά θα βρείτε ο καθένας την αίθουσά του. Δεύτερη πληροφορία. Εφιστώ την προσοχή ε, των Ευρωβουλευτών και των βοηθών τους ότι στην ε, έξοδο της αίθουσας θα σας δοθεί μία κόλλα χαρτί, αυτό το χαρτί συγκεκριμένα, έτσι ώστε να μπορέσετε κι εσείς να δείτε το ωράριο και να κάνετε κάθε φορά να βγάλετε μια φωτογραφία με την εθνική σας αντιπροσωπεία. Είναι σημαντικό για τον τύπο και για όλους τους παρόντες εδώ. Εθνικές αντιπροσωπείες λοιπόν, θα βρείτε στο φάκελό σας μια φωτογραφία με το κοριτσάκι, ένα ωράριο, πότε δηλαδή είναι η στιγμή της χώρας σας. Αριστερά στην έξοδο υπάρχει ένα μεγάλο πανό με το, με το κοριτσάκι και θα πρέπει να βγάλετε όλη φωτογραφία έτσι ώστε στι επόμενε μέρε να μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε, να αποφελθείτε. Τέλο, τώρα, τώρα. Πρώτο εγχείρημα. Καλό του συζητητέ να κατέβουν στην αίθουσα και να πάνε μπροστά από το βήμα. Ταυτόχρονα όλοι όσοι είστε στην αίθουσα θα μαζευτείτε προς το κέντρο της αίθουσας έτσι ώστε ο γεμό να μπορέσει να βγάλει μια φωτογραφία οικογενειακή όλων όσοι είμαστε παρόντες εδώ. Λοιπόν, άρα οι εισηγητέ, παρακαλώ, φύγετε από το βήμα, κατεβείτε και σταθείτε μπροστά από το βήμα. Και εμείς όλοι θα σηκωθούμε και θα κατευθυνθούμε στο κέντρο της αίθουσας για να βγάλουμε φωτογραφία.